E, Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζουμε τη Συνόδο της Ολομέλειας. Τα πρακτικά της χθεσινής ε, συνεδρίασης ε, ε, είναι πλέον προσβάσιμα. Ε, υπάρχουν παρατηρήσει μήπως για τα χθεσινά πρακτικά. Όχι, οπότε θεωρούμε ότι τα χθεσινά πρακτικά εγκρίνονται. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης προβλέπει